συνοπτικά πρακτικά της ε, χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσεις, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Η ημερήσια διάταξη τώρα